The President! <clears throat> Συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Πρώτα απ' όλα, έχω μια ανακοίνωση να σας κάνω, η οποία αφορά μια γραπτή δήλωση, την γραπτή δήλωση υπαριθμών 22, ε, που έχει υποβληθεί από τους Γκέι Μίτσελ, Νιρς Ντέβα, Μάριαν Χάρκιν, Πίτερ Σκίνερ και Αντζέλικα Βέρτμαν ε, σχετικά με την επιληψία. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι έχει υπογραφεί από την πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και σύμφωνα με τον ε, κανονισμό 123 θα διαβιβαστεί δεόντως ε, και θα δημοσιευτεί στα πρακτικά των εγκεκριμένων κειμένων της σημερινής Ολομέλειας και τα ονόματα των υπογραφών των θα δημοσιευτούν στα πρακτικά. Κυρία Βέρτμαν. εξ ονόματος ε, της ε, ομάδας εργασίας ε, για την επιληψία και εξ ονόματος των συναδέλφων Μίτσελ, Ντέβα, Χάρκιν και Σκίνερ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους υπέγραψαν την γραπτή μας δήλωση υπ. 22. 440 υπογραφές έχουμε λάβει και ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα πείσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να βοηθήσει τα 6 εκατομμύρια ανθρώπων. Ευχαριστώ όλους λοιπόν ε, για την στήριξή τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος και συγχαρητήρια σε όλους τους ε, συγγραφείς της δήλωσης αυτής. Νομίζω ότι θέλει το λόγο ο κύριος Εμάνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ε, έχουμε έναν ιδιαίτερο ε, καλεσμένο, τον Βόλφιο Γιακόβιεφ, ο οποίος ήρθε από την Φάτιμα και